Alors, bonjour. non siamo in molti colleghi, però sono già le 9 e 10 e io farei questa proposta, se siete d'accordo. Per rispettare proprio. Λοιπόν, θα πρέπει να ξεκινήσουμε για να σεβαστούμε λίγο τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ξεκινήσουμε. Πριν τελειώσουμε πριν από τις 10 θα διακόψουμε. Έτσι να υπάρξει, θα υπάρξει ένας κενός χρόνος ανάμεσα στη συζήτηση και στην ψηφοφορία. Είναι 9 και 10 όμως και γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε. Κάποιοι συναδελφοί είναι μαζί μας και επαναλαμβάνω αν τυχόν τελειώσουμε νωρίτερα θα σταματήσουμε για όσο χρόνο χρειάζεται. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να σεβόμαστε τους χρόνους. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πρακτικά της επίσκεψης της αντιπροσωπείας της Ήτρες στην Ιρλανδία, 29 μέχρι 31 Οκτωβρίου του 12. Εγώ είμαι η συγγήτρια. Θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση. Ξέρετε ότι υπήρξε αυτή η αντιπροσωπεία. Σε αυτό το ταξίδι λοιπόν πήραν μέρος αρκετοί συνάδελφοι, Ο κυρία Ντελ Καστίγιο, Δε Κάμπος, Κράμερ, Χέλμερ και τα λοιπά. Και ο κύριος Σκέλη ήταν ε, φυσικά ε, λόγω της ε, Παραμονή του στην Ιρλανδία ως Ιρλανδός συνάδελφος, τοπικός συνάδελφος. Συναντήσαμε τους ε, αρμόδιους υπουργούς για τις αρμοδιότητές μας που θα συναντήσουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Δύο από τους υπουργούς λοιπόν συναντήθηκαν μαζί μας και ήταν χθε μαζί μας. Ο ένας είναι ο Πατ Ράμπιτ και ο άλλος ο κύριος Μπρότον e Rabbit per l'energia e le telecomunicazioni. Inoltre durante il nostro viaggio abbiamo, come abbiamo fatto ieri in comunità... όπω είπαμε χθε λοιπόν και χτες, προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε λίγο την πραγματικότητα στην οποία ζει η Ιρλανδία σήμερα. Είχαμε ως συνήθως μια ιδιαίτερα βεβαρημένη μερίσια διάταξη, συναντηθήκαμε με αρνητές του Royal College, εκπροσώπους της αρχής για τις αηφόρες πηγές ενέργειας, υπεύθυνους για τη βιομηχανία, με την Ιρλανδική εργοδοσία, με βουλευτές της ομολόγου μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, Μας παρουσιάστηκαν και οι προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας, οι οποίες ακούστηκαν και χθες εδώ. Έχει πολύ ενδιαφέρον να κατανοήσει κανείς πως ε, για την Ιρλανδία η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει το βασικό σημείο αναφοράς για την οικονομία τους και πώς έχουν πραγματικά μια ουσιαστική επιθυμία να ενισχύσουν την ενιαία αγορά και τις κοινοτικές πολιτικές. Η Ιρλανδία ζει μια δύσκολη κατάσταση λόγω ακριβώς της κρίσης η οποία υπάρχει Συνεχίζουν να υπογραμμίζουν οι Ιρλανδοί συνάδελφοι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρώπη να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις. Υπογράμμισαν επίσης την μεγάλη σημασία την οποία έχει ο ρόλος ε, στη χώρα τους η έρευνα και η καινοτομία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρώ ότι θα έχουμε συμμάχους τους Ιρλανδούς στην προσπάθεια που έχουμε επανειλημμένα εκφράσει να στηρίξουμε καλύτερα οικονομικά το σύστημα της έρευνας. Σε αυτό πιστεύουμε τα ίδια λοιπόν με τους Ιρλανδούς συνοδοιπόρους μας πλέον. Ένα άλλο θέμα στο οποίο κάνουν μεγάλες προσπάθειες οι Ολλανδοί είναι στις επενδύσεις στις ε, υποδομές και στις ανανεώσιμες πηγές. Και επιμένουν επίσης και στα θέματα της ψηφιακής ε, ατζέντα, όπως λέγεται και χθε μας παρουσίασαν εισαγωγικά και μας μίλησαν και για αυτή την Ολομέλεια του Ιουνίου του 2013 γύρω από το θέμα της ψηφιακής επικαιρότητα. Η Ιρλανδία θα παρουσιάσει σε έφετο χρόνο την γενικότερη στρατηγική της γύρω από τα θέματα αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω μετά από αυτήν την σύντομη αλλά πυκνή αποστολή. Ε, ο κύριος Κέλλη θέλει να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ για την σύντομη παρουσίαση της επίσκεψης ε, της αντιπροσωπείας στο Δουβλίνο. Από εκείνη την περίοδο και μετά μίλησα με συναδέλφους στην Ιρλανδία πράγματι εξετίμησαν δεόντως οι τοπικοί παράγοντες ε, τις προσπάθειες τις οποίες κάναμε και την, την κατανόηση που δείξαμε. γιατί δεν έχουν πολλές φορές τη δυνατότητα να συναντηθούν με ευρωβουλευτές. Λοιπόν, ε, ευχαριστώ κυρίως τους ευρωβουλευτές οι οποίοι πήγαν εκεί. Ήμασταν μια ισχυρή ομάδα, σωστά ενημερωμένη. Η ημερήσια διάταξη ήταν πάρα πολύ πυκνή και έτσι δεν καταφέραμε να δούμε το Δουβλίνο ή να ψωνίσουμε κάποιο αναμνηστικό. Λίγος ελεύθερος χρόνος επιπλέον θα ήταν πολύτιμος για όλους, γιατί το να ξυπνάει κανείς και να αρχίσει τις συνεδριάσεις και να δουλεύει στο βράδυ και μετά να μπαίνει στο αεροπλάνο για να φεύγει είναι λίγο βαρύ είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, αν και είναι παραγωγικό βέβαια. Πάντως ε, έδειξε και την προσπάθεια που κάνουν οι φίλοι της Ιρλανδικής Προεδρίας. Οι προσπάθειες τις οποίες έχουν κάνει οι φίλοι της Προεδρίας μέχρι τώρα ήταν αρκετά χρήσιμες το προσωπικό το οποίο προωθεί ε, κατά κάποιο τρόπο τις προτεραιότητες της Προεδρίας θα παίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και φαίνεται ότι τον παίζει σωστά. Ευχαριστώ λοιπόν για τον τρόπο με τον οποίο προεδρεύσατε και για τη θετική σας στάση η οποία μεταφέρθηκε και σε όλες τις ομάδες τις οποίες συναντήσαμε στο Δουβλίνο. Ευχαριστώ τον κύριο Κέλλη. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Όχι, θα συμφωνήσω και εγώ με τον κύριο Κέλλη και το έλεγα στην Προεδρία, στη Γραμματεία προηγουμένως, ότι στις επόμενες συναντήσεις τις οποίες θα κάνουμε ε, θα ελέγξω λίγο το χρονοδιάγραμμα γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία με να χρησιμοποιούμε πλήρως και απολύτως το χρόνο μας αλλά έχει μεγάλη σημασία να γνωρίσουμε και την πραγματικότητα που επικρατεί στις χώρες αυτές. Να μην έχουμε δηλαδή πάρα πολύ πιεσμένο θα έλεγα χρονοδιάγραμμα, αυτό ε, δεν είναι σωστό. Θέλουμε λίγο μεγαλύτερες ανάσες, σε πάση περιπτώσει. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο θέμα. Είναι η, αντι... η επίσκεψη η αυτή. αντιπροσωπείας στο Πακού. Πιλάρ Καστήλιο. Υπεύθυνη τη αντιπροσωπεία. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να σας ενημερώσω και εγώ, πολύ σύντομα θα ήθελα και εγώ να σας ενημερώσω για αυτή τη διάσκεψη κορυφής για την ε, κοινωνία της πληροφορική που χώρα στο Μπακού 6 με 9 Νοεμβρίου 2012. Όπως ξέρετε, αυτό το φόρουμ για την ε, διακυβέρνηση την ηλεκτρονική και την κοινωνία των ε, πληροφοριών. Έλαβε χώρα για πρώτη φορά στην Ισία το 2005 και με στόχο όλες οι ενδιαφερόμενες ομάδες να αρχίσουν σε ίση βάση διάλογο για την ε, θέματα τα οποία αφορούν τις ε, πολιτική της κάθε χώρας σε σχέση με το ίντερνετ και την διακυβέρνηση. Τελικά, ενώ πολλοί ήθελαν να είναι μέλη της αντιπροσωπείας, τρία μέλη κατορθώσαμε να πάμε στον Πακού, εγώ, η Καθρίν ε, Τροτμάν και η Σαμπίν Βερχάιεν. Και δύο άλλοι συνάδελφοι άλλων επιτροπών πήγαν, τους ε, συναντήσαμε κάποιες φορές σε κάποιες εκδηλώσεις. Τελικά έγιναν μέλος αντιπροσωπείων Μαρία Δεζάκη και η κυρία Άντερς Ντότερ. Πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την έβδομη συνάντηση το θέμα είχε σχέση με την ε, διακυβέρνηση μέσω ίντερνετ τα τέχνικα μέτρα που πρέπει να λάβουμε για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ε, ε, πλαστογράφησης της, ε, στις κοινωνίες μας, άλλα θέματα, μέσα και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο ίντερνετ, θέμα που αφορούν την ασφάλεια, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, και τέτοια παρεμφερή άλλα θέματα. Δεν πρόκειται να σας δώσω λεπτομέρειες για όλα τα εργαστήρια, τις συναντήσεις, τις ε, συνεδριάσεις ολομελίας. Απλώς να πω ότι η αντιπροσωπεία μας ήταν πάρα πολύ δραστήρια. Πήραμε σε κάποιες ε, συναντήσεις ως μέλη του πάνελ ε, συμμετείχαμε με μέλη του πάνελ, είχαμε διμερείς συναντήσεις επίσης και θα πρέπει να πω ότι οι υπηρεσίε της Επιτροπής ήταν πάρα πολύ χρήσιμες, διότι όντως είχαμε εξαιρετική υποστήριξη από την γραμματεία Μελετούμε να έχουμε τους πόρους που διαθέτει εκεί η Επιτροπή. Πρέπει να σας πω ότι ο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικός. Υπήρχαν ε, εκπρόσωποι των κρατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι σημαντικός ο θεσμικός ρόλος και του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Είχαμε και την ε, παρουσία της Επιτρόπου Νέλη Κρός, είχαμε διμερεί συναντήσεις μαζί της και μετά συμμετείχαμε μαζί της όλες αυτές τις μέρες σε διάφορες εκδηλώσεις. Θα πρέπει επίσης να αναφέρω ότι από τις διμερείς συναντήσεις αναφέρω αυτές που είχαμε την ΑΕΚ με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, αλλά θα αναφέρω ιδιαίτερως μία που είχαμε με βουλευτές εθνικών κοινοβουλίων από διάφορες χώρες. Δεν ήταν πάρα πολλοί, πολύ άριθμοι, αλλά επανήλθαμε στο θέμα ότι θα πρέπει να έχουμε μία κοινή προσέγγιση για το θέμα αυτού του φόρουμ της ΑΕΦ. Και στο μέλλον θα πρέπει να ενεργούμε με πιο συντονισμένο τρόπο. Τα πράγματα, όπως όλοι λέμε πολλές φορές γίνεται πιο δύσκολο, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε για να προετοιμαστούμε για την επόμενη συνάντηση πιο έγκαιρα. Θα πρέπει επίσης να αναφέρω κάτι το ιδιαίτερο. Έλαβε χώρα στον Πακού, στο Ζερμπαϊζάν αυτή η συνάντηση. Και η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για αυτό το ειδικό θέμα βεβαίως ήταν τεχνολογία εχμής σε μια χώρα ιδιαίτερη με πολλούς φυσικούς πόρους. Πρόκειται για μια χώρα σε πλήρη φάση ανάπτυξης. Η στάση και η Κάποιες δράσεις της κυβέρνησης του Αζερβαϊτζάν έγιναν αντικείμενο κριτικής από κάποιους ε, δημοσιογράφους, κάποιοι από τους οποίους ε, συνελήφθησαν, διότι μέσω ίντερνετ εξέφρασαν κάποιες απόψεις. Και ήταν κάπως περιορισμένη η ελευθερία έκφρασης. Άρα σε όλο αυτό το θέμα υπήρχε ένα μεγάλο ερωτηματικό. Η Επίτροπος ε, Κρός απεφάσισε το θέμα αυτό να το συζητήσει σε μια ζήτηση τρογγυλής τραπέζης. Και έγινε τελικά μια ανακοίνωση, μια δήλωση της Επιτροπής Και εμείς τα πέντε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογράψαμε. Αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν έγινε αποδεκτή θετικά αυτή η δήλωση από την κυβέρνηση. Και η εντύπωση είναι ότι δεν ακολουθεί πλήρως τους κανόνες τους δημοκρατικούς ως χώρα το Αζερβαϊτζάν. Κάποιες ελευθερίες, όπως η ελευθερία της έκφρασης, είναι κάπως περιορισμένες. Η εμπειρία Λοιπόν, σε κάποια θέμα ήταν καλή, σε κάποια άλλα δημιουργήθηκαν ερωτηματικά. States uh, regarding the um, multi-stakeholder uh, nature. Λοιπόν, κάποιες κυβερνήσεις προσπάθησαν να δώσουν σε αυτή τη συνάντηση IAF ένα τόνο πιο κυβερνητικό. Δηλαδή να έχουν την προσέγγιση bottom up, από κάτω προς τα πάνω. Και πολλοί ανησυχούσαν κατά τη διάρκεια του χρόνου προετοιμασίας, του προηγούμενου χρόνου, μήπως υπήρχε κάποιος κίνδυνος για την IF. Η ΑΕΦ λοιπόν, οι συμμετέχοντες, είπαν ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί αυτή η προσέγγιση. Του χρόνου θα γίνει η επόμενη συνάντηση και θα ήθελα να αναφέρω επίσης ότι και η βεβαίως βοήθησε πάρα πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την οργάνωση Δημερών συναντήσεων και μας προσέφερε και οργανωτική υποστήριξη. Η Κάθριν είναι εδώ, η Κατρίν Τροτμάν δηλαδή, εξαιρετική συνάδελφος και οι άλλοι συνάδελφοι Είμαστε οι τρεις σωματοφύλακες σε αυτή τη συνάντηση κατά κάποιο τρόπο. Και συμμετείχαμε όλοι με τον ίδιο τρόπο σε αυτό το σεμινάριο. Η κυρία Τροτμάν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνεχίζω λοιπόν μετά από την Πιλάρ για να πω ότι όπως παρατηρήσατε συνάδελφοι ήμασταν μια αντιπροσωπεία αποκλειστικά γυναικεία. 100% γυναικεία. Δεν λυπάμαι γι' αυτό, ήμασταν καλές, αποτελεσματικές. Απλά το υπογραμμίζω, γιατί όχι να το λέμε όταν χρειάζεται. Αλλά πέρα από το αστείο του πράγματος, να πω ότι θα πρέπει να προετοιμάσουμε καλύτερα τα πράγματα στις πολιτικές μας ομάδες και σε επίπεδο Προεδρείου και Προέδρου οι αντιπροσωπείας μας για να μπορέσει να είναι πραγματικά παρούσα και να παίξει ρόλο ήταν πάρα πολύ μικρή. Στο παρελθόν σε αντίστοιχες συναντήσεις ήμασταν πέντε και μάλιστα στην αρχή επτά. Τρεις λοιπόν είμαι πολύ μικρός αριθμός. Αναγνωρίζω πλήρως την ανάγκη να εξοικονομηθούν ποσά. Αλλά δεν ε, μιλάμε για... Μιλάμε μάλλον <clears throat> για συναντήσεις που δεν είναι συναντήσεις με αποφάσεις οι οποίες είναι δεσμευτικές και άμεσα εκτελέσιμες. Και γι' αυτό μπορούμε να μοιράσουμε την παρουσία μας στα διάφορα ατελιέ και στις διάφορες ομάδες εργασίας και έτσι μεγιστοποιούμε την δυνατότητα επιρροής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα σώμα το οποίο έχει ξεκινήσει θα έλεγα πρωτοβουλίες για το φόρουμ αυτό και θεωρεί ότι είναι μια στιγμή στην οποία θα πρέπει να επενδύσουμε ε, σε επίπεδο παρουσίας. Επιμείναμε λοιπόν στην ανάγκη για μεγαλύτερη προετοιμασία, καλύτερο συντονισμό και πολιτικές συζητήσεις για τις ευρωπαϊκές προκλήσεις και την επικοινωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσω. Υπάρχει ανάγκη να συνυπάρξουν οι προτεραιότητές μας και για την προστασία των ανηλίκων και τα λοιπά. Υπάρχει μια παράδοση θα έλεγα γραπτού δικαίου μέσω οδηγιών, μέσω συμβάσεων και είναι βασικό πλεονέκτημα αυτό σε επίπεδο διεθνές, αυτό το γραπτό δίκαιο το οποίο έχει διαμορφωθεί. Είναι θέμα επίσης εξουσίας, είναι θέμα το οποίο θα συζητηθεί ιδιαίτερα στο φόρουμ αυτό που εξαρτάται από τα Ηνωμένα Έθνη. Για το πού τώρα, για τον τόπο, θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε την Ιρλανδική Προεδρία έτσι ώστε οι χώρες μας που είναι μέλη των Ηνωμένων Εθνών να παίρνουν θέσεις στο θέμα του τόπου που γίνονται οι συναντήσεις αυτές ε, που να μην είναι τόσο ε, ε, θα έλεγα παθητικές και για την ελευθερία του λόγου και για την ελευθερία συνάντησης με την κοινωνία των πολιτών είναι παράδεκτο, απαράδεκτο να μας κατηγορούν <clears throat> άσχετα με το τη θέση που πήρε η Νέλη που ήταν καλή και θαραλέα θέση μας κατηγορούν γιατί πήγαμε εκεί, εμείς τη δουλειά μας κάναμε. Αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχουν εκεί ε, ε, ε, μυστικοί αστυνομικοί οι οποίοι παρουσιάζονται σαν εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Τα είχαμε ζήσει παλιά αυτά και στην Τινησία. Και να βλέπει κανείς ολόκληρα ολόκληρες γειτονιές κατασκευασμένες σαν σκηνικό, ε, χωρίς κανέναν άνθρωπο μέσα, μόνο και μόνο ένα σκηνικό για να κάνουν φιγούρα. Ήταν απογοητευτικό αυτό. Είχαν οργανώσει την πόλη για να μην συναντηθούμε με τον πληθυσμό της. Με τον φτωχό ιδιαίτερα πληθυσμό, τον πληθυσμό που δεν έχει καμία σχέση με τα έσοδα του πετρελαίου. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ενοχλητικό και αυτό δημιουργεί προβλήματα στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στο ίντερνετ, το οποίο όλοι επιδιώκουμε. Μετά, ICAN και ITU. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι και εγώ ε, είδαμε ότι το ICAN ακολουθούσε μια κατεύθυνση πιο σοβαρή, πιο δεκτική, που πράγματι ακούει περισσότερο ε, τις ευρωπαϊκές θέσεις και σέβεται το ρόλο μας. Αυτό είναι θετικό. Απ' την άλλη το ICANN δεν έχει τις ευθύνε τις οποίες έχει, θα έπρεπε ίσως να έχει για τη διαχείριση του διαδικτύου. Και υπάρχει από τη μία η Διεθνής Διάσκεψη για τις Τηλεπικοινωνίες, η ITU, και από την άλλη το ICANN. και μεταξύ τους αμφισβητούν θα έλεγα την βασική ε, θα έλεγα αρμοδιότητα. Η ITU είναι απόλυτα διεθνής ε, ε, υπηρεσία και έχει ένα κάποιο πλεονέκτημα. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε περί τίνος πρόκειται. Υπάρχουν πολλές διασκέψεις την επόμενη περίοδο στον τομέα της ασφάλειας και της χρήσης του φάσματος Υπάρχουν πάρα πολλά πρακτικά τα θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν στην Ευρώπη και εμπλεκόμεθα άμεσα. Έχουμε ανάγκη όμως. Αυτοί οι οποίοι κατέχουν τα τεχνολογικά μέσα με τον ένα τρόπο ή τον άλλο να ελέγχουν απόλυτα την κυκλοφορία της πληροφορίας. Και γι' αυτό η ICAN έχουμε συμφέρον να είναι βασικός συνομιλητής οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν βοήθησαν πάντα. Συναντηθήκαμε και με τον πρέσβη τον ΗΠΑ. Έχουμε πολύ καλές επαφές με τον πρέσβη τον ΗΠΑ στον ΆΙΚΑΝ που προσπαθεί να φέρει τις θέσεις μας κοντά. Αλλά για μια ακόμη φορά δεν υπήρξαν συνάδελφοι από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Ε, συναντηθήκαμε με βουλευτές από διάφορες χώρες, αλλά όχι από την μεγάλη αυτή χώρα που έχει μια συμφωνία υπογράψει με τη ICAN και ε, ε, ε, δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του σε σχέση με τους σερβερ πηγής, τους βασικούς, εν πάση περιπτώσει, σερβερς. Υπάρχουν λοιπόν πολιτικά θέματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο συζήτησης θα πρέπει η Επιτροπή μας ε, να συναντηθεί με τους εκπροσώπους του ΆΙΚΑΝ όταν έρθουν στις Βρυξέλλες για να δούμε ποιες είναι οι προοπτικές τους και να είμαστε προσεκτικοί για τις επόμενες διασκέψεις του ITU γιατί θα αποφασιστούν πράγματα που θα επηρεάσουν τις πολιτικές μας και τα οράματά μας σε σχέση με την λεγόμενη ουδετερότητα του διαδικτύου. Τίποτα άλλο, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Λάγκεν. Ευχαριστώ. Σύντομα μια παρουσίαση, μια παρατήρηση μάλλον για τα όσα είπαμε για το ταξίδι της Επιτροπής στο Δουβλίνο. Ε, ήταν καλό το ταξίδι αυτό. Η πειθαρχία των παρόντων δεν ήταν πολύ καλή. Κατά τα λοιπά ήταν πολύ καλή προετοιμασία ε, και από τον συνάδελφο Κέλλη έκανε πολύ καλή δουλειά. Αλλά Υπάρχουν κάποια ερωτήματα που τίθενται. Ε, η συνάδελφος ε, Πιλάρδο Καστίγιο ε, έπρεπε να εκπροσωπήσει κάποιους συναδέλφους στις συναντήσεις με τους υπουργούς. Αυτό δεν είναι σωστό. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο ε, στο τέλος ε, κάθεται, βρίσκεται μόνο ένας ο οποίος είναι παρόν από την ομάδα και όλοι οι υπόλοιποι είναι κάπου αλλού. Δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι καν δίκαιο. εγώ πέταξα στην επιστροφή μαζί με την ε, πρόεδρο. Όταν έχουμε όμως μια τέτοια αντιπροσωπεία που κάνει ένα τέτοιο ταξίδι, ε, πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες και να κάνουμε τις δραστηριότητε που έχουμε οργανώσει. Αλλιώς τίθεται σε αμφισβήτηση η αξιοπιστία μας. Δεύτερον, ε, οργανωτικά θέματα. επί της ουσίας ήταν καλό το πρόγραμμα, ήταν πολύ ενδιαφέρον, αλλά το γεγονός είναι ότι αυτοί οι ιστορικοί κανόνες που έχουμε για ότι οι βουλευτές δεν καταγράφουν την παρουσίασή τους ούτε σε, μια, έναν κατάλογο ας παρουσιών, εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο. Οπότε καλό θα ήταν ε, σε ε, συνεννόηση με τον συνάδελφο Κέλλη να το δούμε ίσω το θέμα αυτό, γιατί δεν μπορούσε ο ίδιο καν να καταγράψει ότι ήταν παρόν, ενώ είχε κάνει ένα ταξίδι 400 περίπου χιλιόμετρων για να φτάσει. Και επίση για του διαρμηνείς. Εκτιμώ πραγματικά την ε, δουλειά του και χαίρομαι πολύ που μου επιτρέπουν να μιλάω τη μητρική μου γλώσσα, αλλά το γεγονό ότι την πρώτη μέρα είχαμε ένα πρόγραμμα 8 ωρών και πάνω και τη δεύτερη μέρα είχαμε μικρότερο, πιο σύντομο πρόγραμμα, αλλά που χρειαζόταν παρόλα αυτά δύο πλήρεις ομάδες για τέσσερις ε, διερμηνείς δηλαδή που θέλαμε Ιταλικά-Αγγλικά, νομίζω ότι αυτό αποτελεί και ε, δαπάνη χρημάτων χωρίς λόγο και οργανωτικά δεν είναι καλό. Ζητήθηκαν... Ε, ζητήθηκε η διερμηνία νομίζω χωρίς να έχει γίνει καλή οργάνωση. Δεν γίνεται αυτό να οδηγεί αυτόματα στο ότι στο τέλος ε, της συζήτησης ε, να είναι οι περισσότεροι διερμηνείς με στις καμπίνες από τους βουλευτές κάτω στην αίθουσα. Οπότε ίσως να πρέπει αυτό να το δούμε για τις επόμενες φορές. Προφανώς δεν έχετε όλη την ίδια άποψη με μένα, αλλά εγώ όπου ήτανε, ε, όπου, όπου έχω πάει, νομίζω ήταν η πρώτη φορά που συνάντησα κάτι τέτοιο τα τελευταία πόσα χρόνια. Επίσης κάναμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις με πολύ διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων, με επιχειρήσεις κτλ. Ένα είναι το συμπέρασμα που βγαίνει. Ότι οι 10 μεγάλες εταιρείες που παρέχουν ε, ε, ίντερνετ, υπηρεσίες ε, ίντερνετ έχουν την έδρα τους στο Δουβλίνο. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε, αν κατάλαβα καλά και από τις συζητήσεις βέβαια που κάναμε με τους προσώπους των ε, εταιριών αυτών, πρέπει να συζητήσουμε τι γίνεται με τους φορολογικούς συντελεστές. Και όταν ε, εκπονούμε διάφορα προγράμματα διάσωσης για συγκεκριμένα κράτη, στην ε, Κύπρο πάλι θα μας προκύψει κάτι παρόμοιο, νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να απαιτήσουν τέτοια, τέτοιες ε, τεράστιες ε, στρεβλώσεις του διαγωνισμού να εξετάζονται. Εντάξει, το φορολογικό δίκαιο είναι δίκαιο εθνικό, <laughs> αλλά δεν γίνεται από τη μία και το Google ας πούμε να έχει 4.500 θέσεις εργασίας στο Δουβλίνο από όλο τον κόσμο ναι, και μιλούμε για 15% μόνο Ιρλανδούς πολίτες, όλοι οι υπόλοιποι είναι εργαζόμενοι από άλλες χώρες και μας το είπαν και άλλοι εκπρόσωποι των ε, ε, εταιριών αυτών ε, μας είπαν ότι είναι στην Ιρλανδία λόγω ακριβώς των ε, πολύ συμφέρουσων φορολογικών συνθήκων που επικρατούν στη χώρα. Αυτό είναι που λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Ζόμπιχ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η επίσκεψη στην Ιρλανδία νομίζω ότι έδειξε και νέε ε, διαστάσεις. Ε, Όντω η επίσκεψη στην Google ε, ήταν πραγματικά πολύ ανακουφιστική, αν δει κανεί με πόσο τεράστια λεπτομέρεια όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι συλλέγουν προληροφορίε, τι αναλύουν και τι παρέχουν σε όλου του χρήστε παντού. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε εμεί τα δίκτυά μα. και από την άλλη Βεβαίω η κοινωνία της γνώσης στην ε, Ευρώπη ενισχύεται σημαντικά. Σε πολύ ε, σύντομο διάστημα έχουμε ε, την δυνατότητα να κάνουμε τεράστιες έρευνες και γενικώ όλο, το, όλο το περιβάλλον εκεί είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία προωθούνται, συγκεκριμένες ιδέες τα κοινωνικά δίκτυα, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ασφάλεια. κατά τη διάρκεια της Ελληνικής ε, Προεδρίας λοιπόν νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ε, σημαντικό σημείο ανάπτυξης γιατί αυτή όντως η ε, επίσκεψη μας έδωσε πολλά, πολλές πληροφορίες και αναγνωρίσαμε ακριβώς αυτή την διάσταση καθώς επίσης και ποιες, ποια θέματα πρέπει και εμείς να αντιμετωπίσουμε ποιες προκλήσεις έχουμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε και είδαμε τι γίνεται και σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν είναι πάντα οι κατάλληλες. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι σύντομες, οι νέοι δεν έχουν ούτε την όρεξη ούτε την, το χρόνο να κάθονται να διαβάζουν τεράστιες σελίδες στο ίντερνετ. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε τι ζητούν οι χρήστες και Βεβαίω θα πρέπει αυτό να γίνει μέσα σε ένα σωστό νομικό πλαίσιο, τουλάχιστον για το μέλλον, έτσι ώστε και οι, α, ε, καταναλωτές να μπορούν να προστατευτούν από περιπτώσεις πατών ή οτιδήποτε. Πρέπει λοιπόν ε, με όλους αυτούς τους ε, νέους, ε, όλους τους νέους τομείς να τους αναπτύξουμε γιατί μπορεί να όντω να αποτελέσουν ευκαιρία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το ταξίδι λοιπόν στην Ιρλανδία ήταν για μένα ένα πάρα πολύ σημαντικό και μας έδωσε εμπειρία την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Grazie. Ancora. <laughs> Excusez-moi, Madame la Présidente, j'ai juste... Euh, Ξέχασα κάτι το οποίο είναι σημαντικό για την Επιτροπή μας. Το ότι δυσκολευτήκαμε να κινητοποιήσουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να για να ήσαν παρούσες. Ε, πρέπει να μας απασχολήσει αυτό. Να πω επίσης ότι είχαμε ένα φύλακα άγγελο που βρίσκεται ε, στο βήμα, Πρόεδρε η συνεργάτης του Κοινοβουλίου, η οποία ήταν εξαιρετική, αξιόπιστη και αποτελεσματική. Πρέπει να το πω αυτό, γιατί σίγουρα η Επιτροπή μας βοηθάει πάρα πολύ όταν πηγαίνουμε σε τέτοιες συναντήσεις. Είχαμε όμως και μια καταπληκτική και φιλική στήριξη από πλευράς Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Και είναι και αυτή η γυναίκα, λέει η πρόεδρος. Κοιτάξτε, έχουμε αλλάξει λίγο τη σειρά. Είχαμε κάποιο χρόνο. Έχει κλείσει η συζήτηση για την Ιρλανδία. Συζητάμε τώρα την αντιπροσωπεία στο Αζερβαϊτζάν. Υπήρξαν κάποιες, αν θέλετε, επιστροφές στα θέματα, αλλά να πω ότι για το Αζερβαϊτζάν λαμβάνουμε υπόψη λοιπόν τα χαρακτηριστικά που είχε η αποστολή αυτή. Έχουμε την αίσθηση ότι τα πράγματα πήγαν καλά, έγιναν κάποιες προτάσεις για καλύτερα να πάνε στο μέλλον. Για την Ιρλανδία ο κύριος Λάγκεν έκανε κάποιες διευκρινήσεις, υπογράμμισε και κάποια θέματα, κάποια προβλήματα που σημειώθηκαν σε αυτήν την αντιπροσωπεία θα το λάβουμε εν μέρη στο βαθμό που εξαρτώνται από εμά τα πράγματα, γιατί κάποια πράγματα εξαρτώνται από εμά, αλλά από τον κανονισμό του Κοινοβουλίου. Πάντως κάθε αντιπροσωπεία πέρα από το περιεχόμενο, από την ουσία θα πρέπει να προσπαθήσει να βελτιώνεται σε σχέση με το παρελθόν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους λίγα λεπτά ακόμα να σας ενημερώσω σύντομα για τη συνάντηση τη χθεσινή των συντονιστών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής εγκρίναμε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος λόγω των αποφάσεων που ελήφθησαν στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα. Η τροποποίηση αφορά την Τετάρτη 18, 18 Σεπτεμβρίου εμείς είχαμε ανάμεσα στις 18 και 19 συνεδρίαση, αλλά παραμένει μόνο η 18. Έχει διαγραφεί η 19 και προστίθεται και η Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου από τις 9 μέχρι τις 12.30, ε, 26 ε, του μηνός και η Δευτέρα ε, επίσης 17 Οκτωβρίου από τις 9 λέει η πρόεδρος θα γνωστοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα αυτό. Θα γίνουν κάποιες εργασίες ε, σχετικά και με τα θέματα των μελετών. υπήρξε μια πρόσκληση από Πλευρά Ελβετίας ε, για τις 27 και 28 Μαρτίου σε αποστολή εκεί, αλλά θα πρέπει να τα καλύψετε τα έξοδα από τον φάκελό σας. Και από το ΕΛΚ <clears throat> τίθεται το θέμα της έκθεσης Ήλιτς, Κάρστ 2020, και θα συζητήσουμε στην επόμενη ευκαιρία που θα έχουμε το θέμα και της ψηφιακής ατζέντα σχετικά με το ε, με επιχειρηματικότητα 2020 <clears throat> το θέμα αυτό έχει μετατραπεί σε έκθεση, σε ψήφισμα μάλλον, και θα αποφασιστεί ποιος θα το λάβει στην επόμενη ε, συνάντησή μας. Κοιτάξτε, διακόπτουμε τώρα για 10 λεπτά πριν ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες. Δέκα ακριβώς. Παρακαλώ ξεκινάμε πάλι. Bene, cominciamo il voto. Prendete posto. Invito i colleghi a prendere. Καλώ τους συναδέλφους λοιπόν να καθίσουν. risorse si pagano le rinnovabili, si bloccano le rinnovabili. C'è una bella confusione. Le test, oui. Bene, allora proviamo a fare un test. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα έλεγχο παρακαλώ στο σύστημα της ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Votazione aperta. Abbiamo due socialisti di troppo. Έχουμε δύο σοσιαλιστές επιπλέον. Πρέπει να αποφασίσετε ποιοι περισσεύουν. Ancora due socialisti di troppo. Παραμένουν δύο επιπλέον οι σοσιαλιστές. Πρέπει να δείτε ποιοι από τους αναπληρωτές δεν θα ψηφίσουν. Bene, Καλώς λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες μας. Θα ξεκινήσουμε με την έκθεση Τζαβέλα. Compromesso 1, a favore. Πρώτη συμβιβαστική, ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές δεκτή. 15 και 24 από κοινού, ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές δεκτά. 29. 29 υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 29. Ψηφίζεται. Πέρα στις ψηφοφορίες. 32 υπέρ, 24 κατά. Κοιτάξτε, όλος περιέργος το σύστημά μου δεν δούλεψε και γι' αυτό εγώ ήμουνα υπέρ. Λοιπόν, έτσι και αλλιώς έγινε δεκτή λοιπόν. Και η συμβιβαστική 2. Τροπολογία 40. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ κατά. Αποχές δεκτή. 43 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα της 43 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 43. Τέλος της ψηφοφορίας, 27 υπέρ, 31 κατά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 3α μικρό υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Α. Για μια στιγμή. Για μια στιγμή. Έχετε δίκιο. Θεώρησα δεδομένο ότι έχει τελειώσει η ψηφοφορία της συμβιβαστικής 3α μικρό. Απορρίπτεται. Η 3α μικρό απορρίπτεται λοιπόν. 3α ε, μικρό μπις τώρα. Υπέρ κατά αποχές δεκτό. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για το 3α μικρό μπις. Κάθε αρχή και δύσκολη λέει η Πέρα της ψηφοφορίας 24 κατά 30, 24 υπέρ μάλλον, 30 κατά, απορρίπτεται και αυτή η συμβιβαστική. Απορρίπτεται. Λοιπόν, ψηφίζουμε τώρα την 57. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 57. chiusa. 39 a favore, 19 contro, approvato. Emendamento 50. 59 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ήμκο 5 υπέρ. Α, για μια στιγμή η ΙΜΚΟ 5 έχει και προφορική τροπολογία υπέρ. Α, υπάρχει μια αντίρρηση. Ναι, εγώ έχω αντίρρηση για την προφορική τροπολογία, οπότε θα ψηφιστεί η ΙΜΚΟ 5 χωρίς την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 81 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 82, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 84 υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 84. Ένας από την ΚΟΕ ε, πλεονάζει. Καλώς τέλος της ψηφοφορίας 29 υπέρ, 29 κατά, απορρίπτεται η 84. Ψηφίζουμε τώρα την 87 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 96 υπέρ κατά αποχές από ηλεκτρονικός έλεγχος για την 96 τέλος της ψηφοφορίας 29 υπέρ 30 κατά απορρίπτεται Τροπολογία 100 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν και για την 100. Τέλος της ψηφοφορία 37 υπέρ, 22 κατά δεκτή. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος και εδώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 112 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 112. Πέρας της ψηφοφορία. Δεκτή. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 121 Τέλος. Δεκτή. 123 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 112, Ζητώ συγγνώμη, η γραμματεία μου λέει εδώ ότι δεν ψηφίσαμε το δεύτερο τμήμα της 112 και το δεύτερο τμήμα της 113. Εγώ νομίζω ότι το έχουμε ψηφίσει το δεύτερο τμήμα της 112. Και η κυρία Τόγια λέει ναι το ψηφίσαμε. Κοιτάξτε υπάρχει μια αμφιβολία γιατί η γραμματεία δεν έχει σημειώσει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Θα ψηφίσουμε εκ νέου το δεύτερο τμήμα, τις 12 και τις 13. Όχι, λέγουν οι βουλευτές. 112 Questo non l'abbiamo votato, credimi. Questo l'abbiamo votato e 132. 113. Eh, Presidente, è stato votato 30... Κοιτάξτε, 30 υπέρ 28 κατά, το δεύτερο τμήμα της 112, λέγει ο κύριος Πρόντι. Scusate. Abbiamo risolto il problema. Κοιτάξτε, λύθηκε το πρόβλημα. Το 112 πράγματι ψηφίστηκε και καταπίπτει το 113. Λάγκεν. Ναι, αλλά η συνάδελφο Καρβάγιο ζήτησε, ε, μάλλον είπε ότι, πρέπει να, ότι έκανε λάθο, οπότε πρέπει να γίνεται να διορθωθεί. Στην ε, ε, ε Ολομέλεια επίση γίνεται. Era stato Κοιτάξτε, τέθηκε άσχημα το πρόβλημα. Νομίζω ότι υπόθηκε ότι δεν είχε ψηφιστεί. Όχι ότι η κυρία Καρβάλιο δεν είχε ψηφίσει. Λοιπόν, δεν υπάρχουν προβλήματα και θα ψηφίσουμε εκ νέου το 112 με ηλεκτρονικό τρόπο. I'm so sorry, Mrs. Chair. Λυπάμαι, Πρόεδρε ψηφίσαμε ξεκάθαρα το δεύτερο τμήμα της 112. Και μετά κάποιος από εσά άρχισε να λέει ότι δεν υπήρξε ψηφοφορία. Υπήρξε ψηφοφορία. Καταγράφηκε η ψηφοφορία. Δεν με ενδιαφέρει το πώς ψήφισε ο καθένας. Ψηφίστηκε όμως και συνεχίζουμε. Πρόεδρε, Κοιτάξτε, 30 ψήφισαν υπέρ, 28 ψήφισαν κατά. Ήταν ξεκάθαρη η ψηφοφορία. Τελειώνει λοιπόν το θέμα, δεν θα ξαναψηφίσουμε. Quando si Ότι ψηφίστηκε, ψηφίστηκε. Λοιπόν. Κοιτάξτε, 30 υπέρ 28 κατά αυτό ήταν το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Απλά να λάβετε υπόψη αυτούς οι οποίοι δεν είχαν την κάρτα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το οποίο αποφασίζουμε. Θα πρέπει τώρα να λάβετε υπόψη ότι κάποιοι δεν είχαν την κάρτα τους, λέει η κυρία Γιορντάν. Yeah. Allora, έχει ζητήσει το λόγο. Κοιτάξτε, έχει ληφθεί μια απόφαση η οποία είναι αυστηρά πολιτική. Γιατί ε, ξεκαθαρίστηκε και ζητώ σε γνώμη αν ε, δημιούργησα μια κάποια σύγχυση, αλλά δεν κατάλαβα καλά τις πληροφορίες που μου δόθηκαν Έχουμε ένα πρόβλημα, έχουμε λύσει τα υπόλοιπα. Έχουμε όμως ένα πρόβλημα το οποίο αφορά το δεύτερο τμήμα της 112, το οποίο ψηφίσαμε. Και το αποτέλεσμα ήταν 28 και 30 ψήφοι. 30 υπέρ, αν θυμάμαι καλά λέει πρόεδρος, και 28 κατά. Η συνάδελφος Χιούμπνερ μας είπε και το είχαμε λάβει υπόψη μας, ότι δεν είχε την κάρτα της για να ψηφίσει. Οπότε το αποτέλεσμα είναι κανονικά 30-29. Ως εκεί εντάξει. Αλλά σε αυτή τη φάση παρεμβαίνει η κυρία Καρβάλιο, η συνάδελφος Καρβάλιο. Και λέει λοιπόν και η συνάδελφος κυρία Καρβάλιο ότι ανακοίνωσε στη γραμματεία ότι έκανε λάθος η κυρία Καρβάλιο. Έκανε ένα λάθος η κυρία Καρβάλιο και γι' αυτό ζητάει από εσά, όχι εγώ δεν μπορώ να σας το ζητήσω, ζητάει από εσά να το λάβετε υπόψη σας. Ο κύριος Τούρμες έχει το λόγο, μετά η κυρία Τόγια και μετά θα κλείσουμε. Ο κύριος Τούρμες. Εάν αρχίσουμε να επανεμερχόμαστε σε ψηφοφορίες, διότι κάποιος υπέστη σύγχυση θα ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας. Ψηφίσαμε, ψηφίσαμε, ακόμη και αν κάποιες ομάδες δυστυχώς έχασαν, πρέπει να συνεχίσουμε. Διαφορετικά, πραγματικά, θα δημιουργήσουμε μια κατάσταση την οποία δεν θα μπορείτε κι εσείς να προεδρεύσετε και να προχωρήσουμε και να ψηφίσουμε σωστά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι μπορώ να είμαι όσο περισσότερο διαθέσιμη γίνεται. Σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε για το 112β. Εγώ έδωσα σημασία σε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να πω ότι η ανακοίνωση για λάθη και τέτοια στην ψηφοφορία δεν έγινε αμέσως. Μπορεί κανείς να ξαναψηφίσει να ζητήσει την εκ νέου ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Αυτό το οποίο έγινε τώρα εδώ έγινε πολύ αργότερα. Μετά από μία-δύο ψηφοφορίες ε, ξαφνικά βγαίνει κάποιος και λέει πεντέξι τροπολογίες νωρίτερα ε, έκανα ένα λάθος, παρακαλώ να ξαναψηφίσουμε». Έτσι δεν πάει, δεν γίνεται έτσι. Κυρία Πιλάρου. Νομίζω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό, διότι έχουμε πολλές προφορίες. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο είναι σημαντικό, να λαμβάνεται, να ληφθεί υπόψη το πώς ψήφισε η κυρία Χίμπνερ. Διαφορετικά με ένα ψήφο παραπάνω, με ένα παρακάτω αλλάζουν τα πράγματα για μας. Αυτό είναι πρωταρχική σημασία, να ληφθεί υπόψη το πώς ψήφισε η συνάδελφος. Διότι δεν είχε ληφθεί υπόψη. Τώρα, η κυρία Καρβάλιο. Ας ακολουθηθεί η διαδικασία η συνήθι στην Επιτροπή. Μπορεί να αλλάξει, να ψηφίσει διαφορετικά στην Ολομέλεια. Και ας συνεχίσουμε παρακαλώ, αλλά να ληφθεί εφ' εξής υπόψη ο τρόπος με τον οποίο ψήφισε η κυρία Χίμπνερ. Ευχαριστώ. Ε, Λοιπόν, να κλείσει η συζήτηση αυτή. Α, όχι, κάποιος άλλος έχει στήσει το λόγο. Δεν ξέρω γιατί δεν μου δίνετε το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Εγώ απλώ και μόνο θα ήθελα να κάνω μία υπενθύμηση και να θυμίσω τον εσωτερικό κανονισμό που λέει με σαφήνεια ότι βεβαίω μπορούμε να αλλάξουμε όταν κάνουμε λάθο τον τρόπο που ψηφίζουμε και ότι αυτό δεν έχει επιπτώσει σε μία παρελθούσα ψηφοφορία. Διαφορετικά, αν θέλετε, μπορούμε να ξανακάνουμε όλε τι ψηφοφορίε. Αυτό το λέγει και ο ιστορικό κανονισμό. Μπορεί να το επαληθεύσει η γραμματεία. Μετά μπορούμε να διορθώσουμε αυτό που κάναμε. Αλλά ψηφίσαμε, τελειώσαμε, αναγγείλατε το αποτέλεσμα 30 προ 28. Αν η κυρία Χιούμπνερ δεν έχει την κάρτα τη, εδώ και μισή ώρα ψηφίζουμε. Θα μπορούσε εδώ και ώρα να πάει να βρει την κάρτα τη. Κοιτάξτε, κλείνει το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία είναι αυτή η οποία ανακοινώθηκε, απλά προστίθεται η ψήφος της κυρίας Χιούμπνερ, η οποία πρέπει να στείλει κάποιον να φέρει την κάρτα της. Α, ωραία, της τη την κάρτα της την κυρία Χιούμπνερ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ζητώ συγγνώμη για τη σύγχυση που δημιουργήθηκε, αλλά πραγματικά η ενημέρωση δεν έγινε με τον σωστό τρόπο. Φτάσαμε τώρα στη συμβιβαστική 7. Συμφωνείτε όλοι ελπίζω. Ποιοι είναι υπέρ της 7. Κατά. Αποχές. Δεκτή η 7. Περνάμε τώρα στην 133. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή η 133. Ρέτζι 14 τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ρέτζι 3 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την Regi 3 ένας επιπλέον από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα παρακαλώ. «27 υπέρ 28 κατά απορρίπτεται». Φτάνουμε τώρα στην 136, η οποία όχι έχει καταπέσει 136 και συμβιβαστική 8, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 8α μικρό, υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη συμβιβαστική 8α μικρό. Πέρα της ψηφοφορίας. 28 υπέρ 32 κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 β μικρό υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 150, 199 και 200 από κοινού υπέρ κατά αποχές δεκτές. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. 183 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 190 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 24 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 193 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 196 και εδώ υπάρχει προφορική τροπολογία, είναι κατά. Η συνάδελφος χωρίς προφορική τροπολογία 196 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ρέτζι 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ένβι 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 223 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 100 ή μάλλον 224 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 225 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. 227 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. 229 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 234 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 235 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ρέτζι 17 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 236 υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. 238 και 46 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δε, απορρίπτονται. 239 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 240 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 240 παρακαλώ. Ψηφίζεται. 34 Δεκτή. 241 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 243 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 243. πέρα στις 29 υπέρ 31 κατά απορρίπτεται. 245. 245 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 245 ψηφίζεται. Τέλος της ψηφοφορίας. 27 υπέρ 33 κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 250 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 262 α όχι επανερχόμεθα ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 250 τέλος 24 υπέρ 36 κατά απορρίπτεται 262 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 264 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 265 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Άφετ 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 270 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 13α μικρό υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 135 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Μου φαίνεται δεκτό, αλλά θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για το 135 δεύτερο. Πέρα της ψηφοφορίας. 31 υπέρ 27 κατά δεκτή. Δύο υπέρ κατά αποχές δεκτή. Άφετ 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 288 σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 2.96 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 2.98 υπέρ, προφορική τροπολογία. Κατά, αποχές, δεκτή. Άφετ 12 σε τρία τμήματα. Α, όχι, για μια στιγμή έχει καταπέσει η 12, συγγνώμη. Συμβιβαστική 16, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 308 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 308 ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. 32 υπέρ 29 κατά δεκτή. 310 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 311 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 320 και 321 μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 320 και 321. Ψηφίζουμε. ...35 υπέρ, 25 κατά δεκτή. 3.23 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 3.24 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 3.25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 326 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 338 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 338. πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή 35-25. Συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 340 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 362 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 362. Πέρασε της ψηφοφορίας. 34 υπέρ 26 κατά δεκτή. 366 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Διαδικαστικό έχει ζητήσει ο κύριος Ζαντό το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, η Γραμματεία ίσως μπορεί να μου δώσει μια εξήγηση. Δεν πρόκειται για την τροπολογία που καταθέσαμε, για την φράση την οποία δεν γι' αυτό την αποσύρω, δεδομένου ότι δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο είχα υποβάλει εγώ στην τροπολογία. Λοιπόν, αποσύρατε την τροπολογία σας βασικά η τροπολογία σας καλύπτεται από την συμβιβαστική 22. Όχι, ακούστε. Είχαμε προτείνει πάρα πολλές φορές μια πολύ συγκεκριμένη τροπολογία η οποία είχε ίσως το μειονέκτημα είναι κατά του SSS. Δεν, το, το προτείναμε, ε, δεν την προτείναμε σε την τροπολογία, προτείνεται κάτι διαφορετικό από τη γραμματεία. Αυτό λοιπόν το κομμάτι που ψηφίζεται σήμερα δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο είχαμε καταθέσει εμείς. Γι' αυτό την αποσύρουμε την τροπολογία. Καλώς λοιπόν, 374 υπέρ. 374 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 377 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 377. Πέρα στις ψηφοφορίες. 33 υπέρ 28 κατά δεκτή. 381 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό και το δεύτερο. Συμβιβαστική 23. Α, α όχι, συγγνώμη, διακόπτει η πρόεδρος. 382 πρώτα, 382. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος Πέρας της ψηφοφορίας. 28 υπέρ 32 κατά απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Λοιπόν, συμβιβαστική 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 23α μικρό υπέρ κατά αποχές δεκτή. 390 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 393 υπέρ Α, συγγνώμη, έκανα λάθος, λέει η Πρόεδρος. Κοιτάξτε, θα ψηφίσουμε την 393, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 395, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 405 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 412 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 400 για μια στιγμή 417 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 418 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αφέτ 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αφέτ 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αφέτ 7 υπέρ κατά αποχές Πέρας της ψηφοφορίας. 31 υπέρ, 30 κατά δεκτή. 28 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Αφετ 5 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 427 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Ίνκο 26 καταπίπτει. Συμβιβαστή. Ε, συγγνώμη. 4.28 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 4.29 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 29 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 30 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 403 numéro ναι, ναι. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ξεχάσαμε κάποιες τροπολογίες. Η 443 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 444 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Θέλετε να υπάρξει έλεγχος για την Ήμκο 16. Ψηφίζουμε. prima del compromesso 30. Prima del compromesso di voto sbagliata, non c'è compromesso 30. Eh, Inco 16 se, è davanti al compromesso 30 prima del Λοιπόν, πριν από τη συμβιβαστική 30 υπάρχει η ΙΜΚΟ 16. Δεν το βλέπετε. Δεν είναι στον κατάλογο της κυρίας Τόγια. Κοιτάξτε λίγο γιατί ίσως έχουμε εδώ ε, κάτι το μη κανονικό στον κατάλογο. Θα μας βοηθήσει η σκιώδη συγγήτρια της ομάδας μου. Λοιπόν, ψηφίζουμε τώρα την ΙΜΚΟ 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. 27 υπέρ, 31 κατά, απορρίπτεται. Λοιπόν, το 30 το ψηφίσαμε. Περνάμε τώρα στο 403. 403 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 459 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 460 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 466 σε δύο τμήματα. Α, όχι. Στην 466 μόνο το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, α, ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 466. Ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 32 κατά απορρίπτεται. απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 468 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 486 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 488 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 489, 91 και 92 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. Ήμκο 13 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 493 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 494 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 33 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 520 υπέρ κατά αποχές δεκτή 520, 505 μάλλον υπέρ κατά δεκτή 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή 524 υπέρ κατά αποχές δεκτή ΙΜΚΟ 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ρέτζι 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Άφετ 13 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος για την ΑΦΕΤ 13. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή. ΑΦΕΤ 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος μάλλον για την ΑΦΕΤ 11. Τέλος της ψηφοφορίας. 21 υπέρ, 39 κατά απορρίπτεται. Απορρίπτεται λοιπόν η 11, ΙΜΚΟ 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. ΕΝΒ 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. ΙΜΚΟ 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέτζι 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την Ρέτζι 4. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. 33 υπέρ, 26 κατά δεκτή. Άφετη 14 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Ένβι 26 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Άφετ 18 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Άφετ 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Άφετ 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μετά α, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τελική ψήφος, ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Α, έχει ζητήσει ε, κύριε Μαντουρέλ το λόγο. Μπορείτε να μας δώσετε ένα λεπτό για να μπορέσουμε εμείς στην ομάδα να πάρουμε την οριστική μας απόφαση. Ευχαριστώ. Διακόπτουμε λοιπόν ένα λεπτό, για το ζήτηση η Σοσιαλιστική Ομάδα, λέει ο Πρόεδρος. Possiamo riprendere il voto. Λοιπόν, θα πρέπει να επανέλθουμε στην ψηφοφορία, λέει η Πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία, λοιπόν. Ψηφίζεται. Avete votato tutti? Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίζουμε την έκθεση της κυρίας Τζαβέλα. Ψηφίσατε όλοι, τέλος της ψηφοφορίας. 35 υπέρ, 9 κατά 14 αποχές, γίνεται δεκτή η έκθεση. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. E passiamo al voto successivo che riguarda la risoluzione sullo stress test. Prego. Επόμενη ψηφοφορία, stress test λοιπόν των πυρηνικών μονάδων. Συμβιβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 19, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Ηλεκτρονικός έλεγχος το 19, άρχεται η ψηφοφορία. 31 υπέρ 26 κατά Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 34 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή 36 υπέρ κατά απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 43 σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα... Α, συγγνώμη, πρέπει να ψηφίσουμε και την 42. 42 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Σε τρία τμήματα είπαμε μάλλον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό το πρώτο. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται το τρίτο τμήμα. Α, όχι, ζητείτε τεστ για το δεύτερο τμήμα τη 43. Ψηφίζεται. Τέλος της ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 31 κατά απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά έλεγχος για την 64 ηλεκτρονικός έλεγχος πέρα στις ψηφοφορίες Εξήντα έξι υπέρ κατά αποχές δεκτή ηλεκτρονικός έλεγχος για την 66. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 74. Την 74, το δεύτερο τμήμα λοιπόν, σε δύο τμήματα, υπέρ του πρώτου, κατά, αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 75, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 91 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 96 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 97 υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 96. Ψηφίζουμε την 96. 53 a 3 contro. 53 προς 3. Εγκρίνεται. «97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται». Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος της 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Στην συμβιβαστική 11 αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 29 προς 29. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11α. Υπέρ κατά αποχές. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 30 προς 28. Εγκρίνεται. οι τροπολογίες 104 και 105 μαζί. Α, όχι, όχι, όχι. Καταπίπτουν. Περνούμε στην 112. Υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 12. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 118. υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση στην 118. Αρχίζει η ψηφοφορία, λίγη η ψηφοφορία. 31 προς 29 εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο μέρος 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 130 στο δεύτερο μέρος αρχίζει η ψηφοφορία λίγη ψηφοφορία 28 προς 30 απορρίπτεται «136 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται». «142 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται». Συμβαστική 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 143. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 146. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για αυτή την συμβαστική τροπολογία 17. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 29 προς 31 απορρίπτεται. 17α υπέρ. Ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση κυρίως για τις συμβαστικές τροπολογίες. Είναι καλύτερα, αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 49 προς 9. 156 ε, συγχωριστά δύο μέρη. Το πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 160 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 161 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 2 και 11 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 και 5 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνονται, αλλά θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Τις, την τροπολογία 4 και 5 μαζί. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 33 προς 25 ε, εγκρίνονται. 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 και 7 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 και 13 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται τελική ψηφοφορία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 Ε, να σταματήσουμε, να σταματήσουμε μια στιγμή, να διακόψουμε την ψηφοφορία μια στιγμή, λέει η Πρόεδρος. Διότι η Γραμματεία λέει, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς, ότι δεν ψηφίσαμε την 157, την 158 και την 159. Πρέπει λοιπόν να ψηφίσουμε για αυτές τις τρεις τροπολογίες. Λοιπόν, ας περάσουμε η ψηφοφορία. Το μικρόφωνο παρακαλώ. Πρέπει, πρέπει, πρέπει, λέει η γραμματεία, να τις ψηφίσουμε οπωσδήποτε. Καλώς ψηφίζουμε λοιπόν την 157 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 158 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ψηφίζεται ηλεκτρονικά. C'è un τρόπο; Ένας του Έλκη είναι επιπλέον. Eh, Λοιπόν, C'est bon. Πέρα τη ψηφοφορία 48 υπέρ, 5 κατά, 7 αποχές. Καλώς. Τελειώσαμε λοιπόν την ψηφοφορία. Bene, passiamo all'ultimo voto. λοιπόν φτάνουμε στην τελευταία ψήφο για σήμερα το πρωί. Σόζα Βάγνερ, ο εισηγητής Σόζα Βάγνερ έχει ζητήσει το λόγο. Πριν την ψηφοφορία έχετε το λόγο κύριε Βάγνερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ένα λεπτάκι μόνο για να επιμείνω στο ότι Έχουμε μπροστά μας μία ψηφοφορία και γνωμοδότηση της Επιτροπής μας που έχει σχετική αξία δεδομένου ότι θέλει να αντιμετωπίσει μία προσωρινή αλλά εξωτερική έκτακτη κατάσταση. Διότι γνωρίζω πολύ καλά ότι η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο για αυτά τα δικαιώματα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Το συντομότερο είναι Γιατί ήθελα λοιπόν γι' αυτό να ευχαριστήσω του σκιώδη ηγητέ για την βοήθειά του, να ζητήσω συγγνώμη, διότι δεν μπόρεσα να του δω προσωπικά τον καθένα όπω θα επιθυμούσα αυτή την εβδομάδα, αλλά είχα κάποιε δυσκολίε εξαιτία τη κακοκαιρία. Ε, έφτασα με καθυστέρηση από την Ισπανία εδώ στι Βρυξέλλε. Bene, grazie. Allora, iniziamo il voto. Καλώς λοιπόν, ξεκινάμε την ψηφοφορία. Από κοινού, τροπολογίες 1, 2, 3. Υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Α, ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρα της ψηφοφορίας. 42 υπέρ 18 κατά δεκτή. Bene, allora andiamo Καλώς. Τώρα πάμε απευθεία στην τελική ψήφο. Ένα λεπτό διακοπή παρακαλώ. Χρειαζόμαστε στην πολιτική μας ομάδα πριν από την τελική ψήφο. Καλώς. Μπορούμε να περάσουμε στην τελική ψηφοφορία, παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας από το ΕΛΚ πλεονάζει. Πέρα τη ψηφοφορία 32 υπέρ 14 κατά 11 αποχέ δεκτή. Τέλος της συνεδρίασης. Η επόμενη συνάντησή μας θα είναι 20 Φεβρουαρίου στις 9 το πρωί. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Ε,